Θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά, ο κύριος Μάρτιν. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Θέλω να τονίσω ότι εδώ έχουμε απλώς το εφαλτήριο και όχι το τελικό αποτέλεσμα. Ως Κοινοβούλιο θεσπίσαμε μαζί με την Κομισιόν τρία κριτήρια που θεωρούμε ότι θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν. Θέλουμε καταρχήν η συμφωνία αυτή να είναι συμβατή με τους κανόνες του ΠΟΕ, να είναι δεύτερον φιλική προς την ε, ανάπτυξη και τρίτον να ενθαρρύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση. Και νομίζω ότι το αρχικό μας σημείο κίνηση, το εφαλτήριο όπως είπα, επινυχάνει 1,5 από τους τρεις στόχους. Γίνεται πράγματι Συμβατεί η συμφωνία αυτή με τον ΠΟΕ και είναι πολύ σημαντική για τη συνέχιση της πρόσβασης στην αγορά μετά από την τροποποίηση της οδηγίας για την ε, πρόσβαση στην αγορά γιατί εκπνέουν οι ρυθμίσεις την 1η Οκτωβρίου του 2014 αν δεν υπάρξει κάποια ενδιάμεση ρύθμιση από εμά. <clears throat> Καταφέραμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε το Καμερούν να είναι συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ. Για το δεύτερο ε, στόχο δεν είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες των Καμερούν, αλλά 40% του πληθυσμού του είναι κάτω από το όριο της ένδυας και υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στη χώρα αυτή. Δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα με τη ρύθμισή μας αυτή η κατάσταση, αλλά σίγουρα βελτιώνται οι προσπάθειες που έχουμε κάνει μέσω της συμβασικό τονού να αυξήσουμε τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και να τονώσουμε την ε, ανάπτυξη. Οπότε μπορώ να πω ότι το 50% ισχύει. Εκεί που αποτυγχάνουμε είναι στην έννοια <clears throat> που έχει πάντα υποστηρίξει το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση. Δεν το κάνει αυτό όμως η τωρινή ρύθμιση, γιατί το Καμερούν είναι η μόνη χώρα <clears throat> στην περιοχή αυτή που θέλει να συμμετάσχει και 7 χώρες της περιοχής δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια περιφερειακή συνεργασία. Προφανώς δεν φταίει το Καμερούν, <clears throat> γιατί οι άλλες χώρες δεν βλέπουν να υπάρχει κάποιο συμφέρον για μια περιφερειακή ένωση γιατί ήδη ως ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εποφελούνται ήδη από προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι μια λαθασμένη εκτίμηση. Εμείς δεν έχουμε δει ποια είναι τα αποτελέσματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή την εταιρική σχέση στο μέλλον. Παραδείγματο χάρη το να υπάρχουν κοινοί κανόνε προέλευση σε όλη αυτή την περιοχή και το πώ αυτό θα βοηθήσει την περιφερειακή ολοκλήρωση. Κατά την απόψή μου όμως δεν έχουμε προσφέρει πρόσθετα ωφέλη πέραν της φιλελευθερωποίησης. Δεν έχουμε προωθήσει την ατζέντα του εμπορίου. Δεν έχουμε τονίσει πως αυτή η εταιρική εμπορική σχέση μπορεί να βοηθήσει να αναπτύξει κάποιες πολιτικές που εντάσσονται στη συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕΠ. Το πρόβλημα δεν είναι μονάχα του Καμερούν αλλά και των άλλων χωρών επειδή μα ενδιαφέρει η γενικότερη ανάπτυξη, εγώ προτείνω στο Κοινοβούλιο να δεχτεί αυτή την αρχική συμφωνία. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που δεν είναι θέμα που έχει να κάνει με την εταιρική σχέση αυτή, αλλά έχει σημασία στα πλαίσια της σύμβαση τη Κοτονού. Είναι η κατάσταση των ΛΟΑΔ στο Καμερούν. Η πρόσφατη νομοθεσία που έχει εγκριθεί από το Καμερούν, ιδίω το άρθρο του ποινικού κώδικα, κολλάζει τις ε, σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου με φυλάκιση πολιετή. Είναι ένα από τα πιο σκληρά καθεστώτα στην Αφρική σε ό,τι αφορά την καταδίωξη των ΛΟΑΔ. Πάρα πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν θίξει αυτό το σημείο. Εγώ τονίζω και πάλι, δεν είναι αυτό από μόνο του επαρκή αποχρόν λόγο για να απορρίψουμε την εταιρική οικονομική σχέση, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Σύμβαση Κοτονού έχει και ρήτρε <clears throat> ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επομένω αυτή η πτυχή τη σχέση μα με το Καμερούν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. προ το παρόν εγώ προτείνω να δεχτείτε την ενδιάμεση συμφωνία. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο της Επιτροπής, ο κύριο Πίμπαλξ έχει το λόγο. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Μάρτιν για την ε, επικοδομητική του στάση σε σχέση με την Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με το Καμερούν. Η ενδιάμεση συμφωνία που υπεγράφει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Καμερούν είναι ένα πρώτο βήμα για να δημιουργηθεί μια περιφερειακή εταιρική σχέση εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αφρικής. Χάρη σε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία, το Καμερούν εξασφαλίζει πλήρη πρόσβαση για όλα τα προϊόντα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμιά διακοπή από το 2008. Μετά από τη σύναψη αυτής της ε, διάμεσης συμφωνίας το 2007 υπήρξαν πολλά ωφέλη σε σχέση με το Καμερούν διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της, του Καμερούν. Η πρόσβαση αυτή περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων όπως είναι οι μπανάνες και το αλουμίνιο παραδείγματος χάρη ή προϊόντα τα οποία έχουν περιορισμένο μόνο περιθώριο προτιμήσεων. Με την τωρινή εντολή της Κομισιόν υπήρξε περαιτέρω δραστηριότητα για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας στην Κεντρική Αφρική για ένα πιο πλήρες καθεστώς εταιρική οικονομικής σχέσης. Θέλουμε να πετύχουμε σημαντική πρόοδο του επόμενου μήνες. Όταν κλείσουν οι διαπραγματεύσεις και κυρωθούν, η Περιφερειακή Συμφωνία θα αντικαταστήσει την πρόσωρινη συμφωνία που είναι και το θέμα της συζήτησης και όπως είπε και ο εισηγητής θα είναι ένα πρώτο βήμα, ένα εφαλτήριο για περαιτέρω συμφωνίες. Εμείς συνεχίζουμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ο εισηγητής σας είπε ότι δεν υπήρχε επαρκής ενθάνηση για να προχωρήσουμε. Αλλά εμείς έχουμε υποστηρίξει την υποστήριξη Έχουμε διεπλασιάσει την υποστήριξη για περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η μεγάλη πρόκληση από τη δική μου σκοπιά είναι ότι οι χώρες αυτές της περιοχής βλέπουν προς το παρόν λιγότερη ανάγκη να ενταχθούν σε μια οικονομική εταιρική σχέση και στρέφονται περισσότερο στις ε, εξωτερικές αγορές και όχι στις ενδοαφρικανικές αγορές. Αυτό είναι μια χαμένη ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε μια καλύτερη πρόοδο με μια συμφωνία και έτσι να ενισχύσουμε μηχανισμούς που θα τονώσουν το, το περιφερειακό εμπόριο. Αυτή τη στιγμή οι εμπορικές ροές είναι τέτοιας μορφής που δεν επιτρέπουν τις χώρες αυτές της Κεντρικής Αφρικής να είναι πιο φιλόδοξες. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατικοποίηση. Όλα αυτά είναι θέματα ιδιαίτερης προσοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διάλογο πολιτικής και στην στοχευμένη χρηματοδοτική μας υποστήριξη προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Το θέμα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του τύπου, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία των δικαιωμάτων και των γυναικών και των ΛΟΑΤ είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Υπάρχουν δύο άλλοι προβληματικοί τομείς που είναι τα, το λαθρεμπόριο ανθρωπίνων ατόμων και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα αυτά και ξέρουμε ότι θα πρέπει να βασιστεί η σχέση μας με το Καμερούν σε μια μακροχρόνια ενατένιση των θεμάτων αυτών όσο αναπτύσσεται η εταιρική μας σχέση σε ένα βιώσιμο δρόμο ανάπτυξης που να βασίζεται σε πλήρη εφαρμογή των ερητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία. Ξέρουμε ότι πρέπει να επιταχύνουμε τι διαπραγματεύσει για τι πρόνοιε ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Καμαρούν, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μα εμποδίσει από του από το να υποστηρίξουμε την ενδιάμεση συμφωνία εταιρική οικονομική σχέση με το Καμερούν, γιατί με τον τρόπο αυτό <clears throat> πιστεύω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε έμεσα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καμερούν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου τη Επιτροπή ΔΕΒΕ, η Τζούντι Θεσσαρτσεντίνη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. προτείνω στην Επιτροπή Ανάπτυξης να πρότεινα μάλλον στην Επιτροπή Ανάπτυξη να μην υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Δεν με άκουσαν βέβαια. Τώρα άκουσα τι είπε ο Ντέιβιντ Μάρτιν και είπε γιατί αυτή η διαμεση συμφωνία δεν είναι τέλεια. Άκουσα μετά τον κύριο Πίμπαλξ, ο οποίο είπε ότι πράγματι υπάρχει πολύ λίγο περιφερειακό εμπόριο. Άρα έχω να πω πολύ απλά το εξή. Όλοι γνωρίζουμε γιατί δεν είναι καλή η κατάσταση για το Καμερούν, αλλά αυτό που κάνουμε τελικά είναι ε, να λέμε το ένα και να κάνουμε το άλλο. Διότι το Καμερούν θα ε, μπορούσε να ε, στείλει τα προϊόντα του σε ανταγωνιστική τιμή στην Ευρώπη γιατί ο κανονισμός περί πρόσβαση στην αγορά έχει προσαρμοστεί για να κάνει λίγο πιο δύσκολες τις ε, συνθήκες για τις ε, χώρες τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Ουσιαστικά επιβάλλουμε κάποιες ε, ειδικές απαιτήσεις σε αυτές τις χώρες που μπορεί να φαίνονται σαν αναπτυξιακές συμφωνίες, αλλά δεν είναι ακριβώς και αυτό που ουσιαστικά καθιερώνουν ε, είναι την ελεύθερη διακίνηση των δικών μας ε, προϊόντων. Αυτό δεν είναι καλό για την ανάπτυξη. Uh, Περνάμε στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Δεν βλέπω στην αίθουσα τον κύριο Στάσνη εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ούτε τον κύριο Κορτές Λάστρα, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω τον ε, συνάδελφο Ρίναλντι από το κόμμα των φιλελευθέρων αν είναι έτοιμος να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για όλους τους συναδέλφους. Αυτό είναι ένα μικρό βήμα αλλά ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε την εμπορική μας πολιτική εναντί των χωρών και θέλω να κάνω μια σύντομη σύνοψη των στόχων αυτής της ε, συμφωνίας. Κάναμε μια μεταρρύθμιση για την βοήθεια προς τις χώρες ΑΚΕ με εστίαση στις πιο φτωχές χώρες. Επίσης είπαμε για, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στις ε, χώρες ΑΚΕΣ και έχουμε και επίσης ενδιάμεσες συμφωνίες όπως αυτή με το Καμερούν. Είναι μια σχετικά βραδία διαδικασία γιατί ξεκίνησαμε το 2002 και είμαστε πάντα σε ενδιάμεσο καθεστώς εμπορικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Αλλά εδώ ίσως μπορεί να μας πει και ο Επίτροπος πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να κυρωθεί η συμφωνία με το Καμερούν. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα κινούνται. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια προσπάθεια πειθούς ώστε και οι δύο πλευρές και οι χώρες ΑΚΕ και η Ευρώπη να κατανοήσουν ότι ο δρόμος αυτός δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος θα τροποποιηθεί επειδή περνάμε δύσκολες χρονικές στιγμές. Είναι ο σωστός δρόμος τον 21ο αιώνα που θα πρέπει να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό των σχέσεών μας. Βλέπετε εδώ τι λέει ο τοπικός ε, τύπος στο Καμερών που είναι σκεπτικιστής. Οι ΜΚΟ έχουν μια αρνητική στάση. Οι επιχειρηματίες λένε ότι δεν συμφωνούν ιδιαίτερα. Τα εθνικά κοινοβούλια πολλές φορές δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όλα αυτά δεν μας βοηθούν ιδιαίτερα. Χρειαζόμαστε για αυτό το λόγο να υπάρξει μια καλύτερη πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την κοινή γνώμη. Σεμινάρια με τους δημοσιογράφους, με τις ΜΚΟ, με τους υπόλοιπους εμπλεκομένους που θα είναι και οι δυνητικοί δικαιούχοι ώστε να κατανοήσουν τα ωφέλη που μπορούν να προσποριστούν από αυτή τη συμφωνία. Ως μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ζήτησα από την Επιτροπή μου να οργανώσει μια επαφή με τον τύπο των Βρεξελών που ασχολείται με τα αφρικανικά θέματα για να είναι σαφέστερη ποια είναι η στάση μας για τα ζητήματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να επιμείνουμε έναντι των χωρών που είναι δικαιούχοι <clears throat> για τα μέτρα εφαρμογής που πρέπει να λάβουν σε εσωτερικό επίπεδο πέραν αυτών που ε, περιλαμβάνει η ενδιάμεση συμφωνία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι θα αποκομίσουν καρπούς από αυτήν την συμφωνία. Αυτό σημαίνει όχι μονάχα αντιμετώπιση της ε, διαφθοράς, αλλά και δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος που εξασφαλίζει πιο ισοδίκια κατανομή των πόρων από αυτή τη συμφωνία. Και τώρα, ο κύριος Κορτές ε, Λάστρα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, οι διαπραγματεύσει αυτέ για τη Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση ε, με τι ε, χώρε ΑΚΕ δεν πηγαίνουν προ την κατεύθυνση μετά από έξι χρόνια και ίσως ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ε, σε μια διαδικασία που από την αρχή ε, χαρακτηρίστηκε ότι άφηνε εκτός σημαντικούς φορείς όπως είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα συζητάμε την επικύρωση της συμφωνίας με την Κεντρική Αφρική και στην προκειμένη περίπτωση με το Καμερούν. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε φορά που έρχεται εδώ η Κομισιόν για να συζητήσει τέτοιες συμφωνίες εταιρικής οικονομικής σχέσης μας λέει ότι πρόκειται για την ανάπτυξη για το ελεύθερο εμπόριο Θέλουμε λοιπόν η ε, ε, Κομισιόν και οι χώρες ΑΚΕ να συμμετάσχουν για τη σύναψη, σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη περιφερειακών αναπτυξιακών συμφωνίων που θα προωθήσουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Κέλλερ από την ομάδα των Πρασίνων. Αν δεν λειτουργεί το μικρόφωνο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διπλάνο. Vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Can take another micro on the next seat. Δοκιμάστε ένα άλλο μικρόφωνο. okay. Uh... Λοιπόν, με αυτή την ενδιάμεση συμφωνία αποδυναμώνεται ολόκληρη η κεντρική Αφρική γιατί οι γειτονικέ χώρες ε, τίθενται σε αντιπαράθεση τελικά για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε επίπεδο ενδίας χρειαζόμαστε παραπάνω πράγματα και όχι μόνο χρήμα. Πρέπει να βοηθήσουμε για να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία και αυτό δεν γίνεται με την ενδιάμεση ε, συμφωνία είναι και αντίθετη με άλλες αρχές ουσιαστικά είναι μια και καλυμμένη αν θέλετε ε, βοήθεια για άλλους σκοπούς οι, οι κοινωνικές παραδείγματος χάνει υποχρεώσει των επιχειρήσεων λείπουν από τη συμφωνία αυτά θα πρέπει να θέσουμε σε πρώτο επίπεδο και όχι τα εμπορικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε συνεργασία για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη δεν είναι ε, για το δικό μας το συμφέρον η συμφωνία αυτή δεν θα έπρεπε να είναι ε, εμείς οι πράσινοι το είπαμε και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και το λέμε και εδώ στην Ολομέλεια ζητούμε από όλους τους συναδέλφους να ξανασκεφθούν ποια είναι τα επιχειρήματα που ενισχύουν την άποψη να βοηθηθεί περαιτέρω το Καμερούν δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ποια είναι η θέση της ομάδας μου για τη στρατηγική της Κομισιόν σε σχέση με την εμπορική συμφωνία με τις χώρες, της, ε, χώρες ΑΚΕ. Έχουμε από την αρχή μια επικριτική στάση. Λέτε ότι αυτή η συμφωνία δεν έχει λειτουργήσει. Το Καμερούν είναι αυτή τη στιγμή η μόνη χώρα η οποία μπόρεσε να πιστεί να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Οι άλλες χώρες της Κεντρικής Αφρικής αποφάσισαν ότι αυτή η συμφωνία μόνο μειονεκτήματα θα τους ε, φέρει. Δεν θέλουν να υποχρεωθούν να ανοίξουν πλήρω τι αγορέ του για τις ευρωπαϊκές ε, πολυεθνικέ. Δεν βοηθάει αυτή η συμφωνία την ανταγωνιστικότητα ε, των χωρών αυτών και επομένως και την περιφερειακή ολοκλήρωση, η οποία απειλείται με το γεγονός ότι γίνεται μια συμφωνία μονάχα με μια χώρα. Και ούτως ή άλλως το Καμερούν θα χάσει την ε, πρόσβασή του στην αγορά της Ευρώπης τον Οκτώβριο του 2014 χωρίς αυτή τη συμφωνία. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν προσπαθεί η Κομισιόν να υποχρεώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνενέσει. Η Επιτροπή Ανάπτυξης η ομάδα μου στην Επιτροπή Ανάπτυξη θεωρεί ότι πρέπει να αποσυρθεί αυτή η πρόταση της Κομισιόν γιατί είναι κακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κακή για τι ε, τις αφρικανικές χώρες και ιδιαίτερα για το Καμερούν. Και δεν προωθεί τη συμφωνία και την ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ. το λόγο στον Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στο παρελθόν η προτιμησιακή πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές δεν θεωρούσαμε ότι βοηθούν ιδιαίτερα τις ε, αναπτυξιακές τους προοπτικές. Ε, είδαμε ότι έπρεπε να γίνουν άλλα πράγματα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου βοήθησε στο να υιοθετηθούν άλλες προσεγγίσεις. Τι, το θέμα που συζητούμε ξεκίνησε από την αρχή της δεκαετίας από το 2000, 2002 και δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα. Γι' αυτό βρέθηκε αυτή η ενδιάμεση συμφωνία σαν εφαλτήριο, σαν ενδιάμεσο βήμα ε, για να προσφερθεί προτιμησιακή προσ... πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές. ε, ε μεταξύ των χωρών της περιοχής μόνο το Καμερούν θεώρησε ότι πρέπει να υπογράψει την ενδιάμεση αυτή συμφωνία πράγμα που έγινε το 2007 αλλά η συμφωνία αυτή απαιτεί τώρα έγκριση και από την Εθνική Συνέλευση η ε, Γκαμπόν και το Κόγκο χρησιμοποιούν το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων ε, και η, αυτό δημιουργεί και μόνο αυτές οι χώρες λοιπόν θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμμετάσχουν όμως εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει να έχουμε μια περιφερειακή συμφωνία όχι συμφωνία με μεμονωμένες χώρες της περιφέρειας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες των χωρών της περιοχής αν θέλουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη. Ε, τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Κάσμαν για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον David Μάρτιν για το έργο του, αλλά συμφωνώ και με άλλου ε, που θεωρούν ότι θα υπονομεύσει δυνητικά την περιφερειακή ολοκλήρωση αυτή η συμφωνία που περιορίζεται σε μια μόνο χώρα τη κεντρική Αφρική, αρχικό στόχο όμω ε, των συμφωνιών ε, οικονομική τερική σχέση, είναι να βελτιώνουν την οικονομική ολοκλήρωση. Πώ λοιπόν η σύναψη διμερίου συμφωνία θα προωθήσει τον στόχο αυτό. Επίση, ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλέ φορέ έχουμε ζητήσει ρητρέ ανθρωπινά δικαιώματα να περιλαμβάνονται σε όλε τι ε, συμφωνίε, Το Καμερούν όμω την κοινότητα ΛΟΑΔ την ε, διώκει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο και πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση που προβλέπεται και μέσω του ποινικού δικαίου. Ο εισηγητής λέει να δώσουμε έγκριση για την ενδιάμεση συμφωνία και σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Πάντω επιμένω ότι μια τέτοια ενδιάμεση σήμερα θα πρέπει να είναι ένα εφαλτήριο προ ενισχυμένε διαπραγματεύσει με όλε τι χώρε κεντρική Αφρική και θα πρέπει να καλύπτουν και σημαντικά ζητήματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη και όχι μόνο το εμπόριο. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστούμε ο συνάδελφος Τυρολιάν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο στόχος στην Κεντρική Αφρική είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την περιφερική ολοκλήρωση αυτή η συμφωνία όμως είναι παραπλανητική γιατί τελικά αφορά μονάχα μία χώρα της ε, Κεντρικής Αφρικής. Η σημερινή Γουινέα δεν συμμετέχει πια στις διαπραγματεύσεις και αυτό σημαίνει ότι και οι άλλες χώρες της Κεντρικής Αφρικής δεν θα θελήσουν να υποστηρίξουν μια συμφωνία που εκπροσωπεί μόνο τα συμφέροντα του Καμερούν. Η στάση της Κομισιόν δεν είναι σωστή γιατί ουσιαστικά ενισχύει τις εθνικές στρατηγικές, οδηγεί σε μια εξειδίκευση σε προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας και διατηρεί τις άνισες συνθήκες ανταλλαγής προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν δεν βελτιώνεται η κατάσταση και δεν προωθεί την δυνατότητα να υπάρξουν ε, περιφερειακές συμφωνίες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Οκτωβρίου 2014. Στη διαδικασία Catch the Eye έχω δύο συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο και θα τον δώσω πρώτα στον συνάδελφο Κούτας. Doamnă președinte, Camerun este Το Καμερούν είναι η μόνη χώρα, χώρα στην Κεντρική Αφρική που ε, διαπραγματεύτηκε ενδιαφέρεται για την ε, ενδιάμεση συμφωνία. Όταν δόθηκε από το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου η δυνατότητα ε, ε μόνο το Καμερούν ε, προχώρησε και ε, αυτό δεν νομίζω δεν ε, ε, αντιπροσωπεύει βεβαίως ολόκληρη την Αφρική αλλά οι άλλες χώρες δεν πιστεύουν ότι είναι έτοιμες να υπογράψουν τη συμφωνία αλλά εμείς πιστεύω ότι πρέπει να παροτρύνουμε το Καμερούν να υπογράψει τη συμφωνία ε, Κυρία Πρόεδρε η προσπάθεια εκδημοκρατισμού της Κεντρικής Αφρικής ε, προσπαθεί να συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες η κατάσταση όμως συνεχίζει να είναι επισφαλής υπάρχει φόβος λοιμού δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα αν λοιπόν δεν καταφέρουμε σύντομα να βοηθήσουμε τους πιο φτωχούς τα πράγματα θα κυκλαμωθεί κλιμακωθούν. Είναι ντροπή πραγματικά ε, η κατάσταση που ισχύει στην Κεντρική Αφρική. Υπάρχουν και ε, γραφειοκρατικά εμπόδια, υπάρχουν πολλοί φραγμοί που δεν επιτρέπουν στους παραγωγούς της περιοχής να εκμεταλλευτούν αν θέλετε την παραγωγή τους. Γι' αυτό λοιπόν νομίζουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να διορθωθούν με αυτή τη συμφωνία. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ. Κύριε Πρόεδρε, με βουλευτές, είναι κρίμα που δημιουργείται τέτοιο ζήτημα με τη Συμφωνία τη Οικονομικής Σχέσης. Δεν ξέρω αν μπορώ να γεφυρώσω το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι ε, οι εμπορικοί κανόνες αποφασίζονται από τον ΠΟΕ. Το σύστημα του ΠΟΕ είναι καλό, είναι κακό, εξαρτάται από τον καθένα, αλλά το έχουν αποδεχθεί όλοι οι εταίροι του ΠΟΕ και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, το καλύτερο είναι σίγουρα να συμφωνήσουμε ε, στο γύρο των αναπτυξιακών της Ντόχα. Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις έχουν τελματώσει στην Ντόχα και τώρα έχουμε την εξή κατάσταση. Οι συμφωνίες ε, για συμφωνιστερική σχέση οικονομικής που είχαμε συμφωνήσει με τους εταίρου δεν μπορούμε ε, να τις δεχθούμε πια γιατί δεν συνάδουν με τις αρχές του ΠΟΕ, δεν είναι συμβατές με τον ΠΟΕ. Πρέπει λοιπόν να είναι και νομικά, ε, να είμαστε και νομικά σωστοί. Ε, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Επίσης, ε, οι επενδύσεις είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, αλλά πρέπει να είναι σαφής και νομική κατάσταση και αυτό και για το εμπόριο. Κατά την άποψή μου λοιπόν αυτή η πορεία είναι ρεαλιστική. Καμακάρι να ήταν περιφερειακές οι διαπραγματεύσεις και συμφωνίες θα ήταν το καλύτερο σίγουρα θα γίνονταν ισχυρότεροι και οι εταίροι και θα ήταν καλό να δουν και το εμπόριο ως έναν τρόπο να ε, βρουν μια διέξοδο από την ένδυα. Σίγουρα ε, για το Καμερούν είναι πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Υπάρχουν πολλοί εμπορικοί εταίροι που υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι σημαντικό επίσης να δούμε πώς βλέπουν και οι δικοί μας εταίροι αυτές τις ε, συμφωνίες. Ε, δημοσία είναι αρνητική, κατηδίαν όμως, ε, αν δείτε και τι έγινε στην πρόσφατη υπουργική διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ, εκεί δεν είναι τόσο αρνητική η στάση τους. Κανείς δεν θα επέβαλε μια τέτοια συμφωνία σε έναν εταίρο, αν και αυτός δεν την ήθελε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο που ζητάνε ουσιαστικά είναι περισσότερος χρόνος για να αναπτυχθούν. Το σύστημα, παραλαμβάνω όμως που έχουμε τώρα, δεν είναι συμβατό με το σύστημα του ΠΟΕ. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε. Εγώ περιμένω να μπορέσουμε να έχουμε μια περιφερειακή συμφωνία οικονομικής σχέσης ε, σύντομα. Ελπίζουμε να λάβει σάρκα και ωστά. Έχουμε και την ε, νέα επίτροπο για το εμπόριο στην Αφρικανική, Κοινότητα, η οποία, ε, Αφρικανική Ένωση, η οποία μας εξέφρασε ακριβώς τις ανησυχίες. Και πρώτη φορά τις άκουσα για να σας πω την αλήθεια. Πάντα λέω στους εταίρους μας, πείτε μας τι δεν σας αρέσει, τι θέλετε να αλλάξουμε. Φυσικά και δεν θα ήθελα συμφωνία που θα έπληκε την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Πάντως ε, πιστεύω ειλικρινά ότι δεν θα πλήξει την ανάπτυξη του Καμερούν αυτή η συμφωνία και ε, το αντίθετο μάλιστα, ότι θα τη βοηθήσει πιστεύω και είναι κρίμα τελικά να έχει δαιμονοποιηθεί και το όνομα ακόμα αυτή τη συμφωνία. Να θεωρείται δηλαδή ότι θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι στι χώρε. Όχι, το αντίθετο συμβαίνει. Εμεί θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη όσο περισσότερο μπορούμε στο διεθνέ εμπορικό σύστημα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε. Πρωτού ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας, θα ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Στάσνη να λάβει το λόγο για δύο λεπτά εάν σύμφωνη και ο εισηγητής. Δεν είναι φυσιολογική διαδικασία. Κύριε Στάσιν, κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ ιδιαίτερα την χειρονομία σας και ε, ζητώ συγγνώμη γιατί θα ερχόμουν νωρίς αλλά δεν τα κατάφερα. Ε, είχα ένα πρόβλημα. Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικού χαρακτήρα είναι ένα πρώτο βήμα για μεγαλύτερη περιφερειακή συμφωνία η οποία θα οδηγήσει σε περιφερειακή ολοκλήρωση όλη τη περιοχή τη Κεντρική Αφρικής. Εγώ υποστηρίζω αυτή τη συμφωνία γιατί θα δώσει ένα μήνυμα για τη συμφωνία της εμπορικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Αφρική. Η οικονομική αυτή εταιρική σχέση μπορεί να γίνει πραγματικός καταλήτης για μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Κεντρική Αφρικής των οικονομιών της περιοχή με ωφέλη για όλες τις περιοχές αλλά μια υπηρετική περιοχή ελευθέρου εμπορίου μπορεί να γίνει εάν συνεχίσει η υπεραιτέρω ολοκλήρωση σε περιφερειακό επίπεδο στην Αφρική. Είναι σαφές ότι οι τωρινές προσπάθειες προς οικονομική ολοκλήρωση είναι ανεπαρκείς και θα πρέπει να εντατικοποιηθούν. Οι χώρες της Κεντρικής Αφρικής θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη προσήλωση στο στόχο αυτό με το να κλείσουν τις διαπραγματεύσεις γιατί η έλλειψη περιφερειακής ολοκλήρωσης είναι πραγματικά ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη που ξεκινάει από το εμπόριο. Είναι πολύ μικρό το ενδοκέντρο αφρικανικό εμπόριο, επομένως η μείωση των ε, φραγμών στον εσωτερικό αυτό χώρο πρέπει να παραμείνει μια προτεραιότητα. Εμείς θεωρούμε ότι το Καμερούν θα είναι μια αναδυόμενη οικονομία μέχρι το 2035, είναι ένας κέριος εταίρος μας στην Κεντρική Αφρική. Ζητάμε από το Καμερούν μαζί με την Καμπόν και την Ισημενή Γουινέα να παίξουν το ρόλο κινητήριας δύναμης για να υπάρξει περαιτέρω περιφερειακή ολοκλήρωση και μια ουσιαστική τελωνιακή ένωση στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής μας David Μάρτιν τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να πω στους συναδέλφους που εξέφρασαν δισταγμούς ε, αν δεν επρόκειτο για ενδιάμεση συμφωνία δεν, θα συμφωνούσα μαζί τους αλλά πρόκειται για ενδιάμεση συμφωνία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει στην πλήρη ολοκλήρωση ήρθε στην Επιτροπή Εμπορίου ο πρέσβης του Καμερούν μας εξήγησε ορισμένα πράγματα και ήρθα και εγώ ε, σε επαφή με τον Υπουργό Εμπορίου που τόνισε τη σημασία της συμφωνίας αυτή για τη χώρα του δεν, χρειάζεται, μπορούμε να τιμωρήσουμε το Καμερούν επειδή δεν είναι λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα όταν όλες οι άλλες χώρες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες δεν δώσουμε περισσότερο σε όλες τις άλλες χώρες με μεγάλη χαρά άκουσα τον ε, ε Επίτροπο να λέει ότι δίνονται περισσότερα κονδύλια για την ενίσχυση περιφερειακών ενωτήτων ε, ναι, στην Αφρική και αλλού πραγματικά λοιπόν ε, θα έπρεπε να ε, είχε γίνει ε, ε, αυτό από πιο παλιά. Δεν το κάναμε πιο παλιά, άρα τώρα έχουμε την ευθύνη να διορθώσουμε τις ζημιές, αν μπορώ να το πω έτσι. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι το εξή. Ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω τη συμφωνία αυτή είναι επειδή πιστεύουμε, πιστεύω ότι ακόμη και αυτά που που προσφέρουμε με τη συμφωνία αυτή ακόμη δεν είναι αρκετά αλλά είναι καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαν οι χώρες αυτές να πάρουν από αλλού. Πιστεύουμε ότι δεν, ε, το 80% που αναφέρεται εδώ είναι ε, καλό όπως υπάρχουν όμως και τα συνοδευτικά μέτρα και γι' αυτό θα ήθελα να την υποστηρίξουμε τη συμφωνία. Ευχαριστώ Πολύ, κύριε Μάρτιν. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έληξε η συζήτηση και η ψηφοφορία για την έκθεση του συναδέλφου Μάρτιν θα διεξαχθεί σήμερα στι 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του συναδέλφου Ιβάη Κάλφιν, περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Θέλω πρώτα απ' όλα να παρακαλέσω τον εισηγητή να πάρει το λόγο ο συνάδελφος Κάλφιν.